το τελικό σχέδιο της ε, ημερησίας διατάξεως που εγκρίθηκε στις 8 Ιανουαρίου από τη διάσκεψη των Προέδρων σας έχει διανεμηθεί. Σήμερα Δευτέρα και επειδή η κυρία Αντρικένε δεν μπορεί να είναι δυστυχώς παρούσα σήμερα το βράδυ για να παρουσιάσει την έκθεσή της για την ανάπτυξη του ε, Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών θα γίνει η συζήτηση αυτή την Τετάρτη και θα ψηφιστεί την Τετάρτη. Για την Τρίτη δεν υπάρχουν ε, τροποποίησεις. Για την Τετάρτη η ομάδα των Πρασίνων ζητεί να, γίνουν, να κατατεθούν και ψηφίσματα μετά από την συζήτηση για την κατάσταση στην Γάζα. Επομένω να είναι συζήτηση με ψήφισμα. Τον λόγο έχει ο κ. Κον Μπέντιτ. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι γνωστή η κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα. Είναι φυσικό να το συζητήσουμε το θέμα στο Κοινοβούλιο. Θα θέλαμε όμως το Συμβούλιο Ασφαλείας να λάβει θέση. Απαιτούμε όλες οι αρχές να λάβουν θέση, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητήσουμε και δεν θα λάβουμε θέση. Νομίζω ότι αν λάβουμε υπόψη τον ε, κατεπίνοντα χαρακτήρα της κατάστασης θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει θέση και να πει τι ακριβώς επιθυμεί για να σταματήσουν οι σφαγές στη Μέση Ανατολή. Είναι απαράδεκτο το Κοινοβούλιο να μην έχει το θάρρος και τη διάβια να ψηφίσει μια πρόταση ψηφίσματος μετά από τη συζήτηση. Γι' αυτό η ομάδα μας θα ήθελε να αναθεωρήσουμε την απόφαση της διάσκεψης Προέδρων και να λήξει η συζήτηση η οποία θα γίνει και πρέπει να γίνει για την κατάσταση στη Γάζα με ένα ψήφισμα το οποίο θα καταδεικνύει τη σαφή και σταθερή θέση αυτού του Κοινοβουλίου με μια, μια πλειοψηφία για να σταματήσουν οι σφαγές στη Γάζα. Θέλουμε, απαιτούμε ένα ψήφισμα, διότι φέρουμε πολιτική ευθύνη έναντι των τεκτενομένων και δεν μπορεί να γίνει μια απλή συζήτηση. Θα πρέπει να κατακυρωθεί από ένα ψήφισμα για να δείξουμε ακριβώς τι καταγγέλουμε, τι επιθυμούμε και τι καταγγέλουμε. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Θα μιλήσει, ο κύριος Σβόμποντα επιθυμεί και ο κύριος Βίρτς να μιλήσει υπέρ της προτάσεως αυτής, αλλά βέβαια μόνο ένας μπορεί να λάβει το λόγο. Σκεφτήκαμε καλά την υπόθεση Με το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών νομίζω έχουμε μια βάση όπου μπορούμε να πούμε και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υποστηρίζουμε το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και όπως είπε και ο ίδιο ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου μπορούμε να ζητήσουμε και από τις δύο πλευρές να θέσουν τα όπλα παραπόδα και να ανταποκριθούν στα κελεύσματα της, ε, του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υπό την έννοια αυτή μπορούμε να δεχθούμε ένα κείμενο ψηφίσματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εφόσον θα απηχεί τα ίδια αυτά πράγματα του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ευχαριστώ. Αντίθετος, ο κύριος Έλμαρ Μπρόκ θα μιλήσει κατά της ιδέας του ψηφίσματος. Νομίζω ότι η απόφαση της διασκέψεως των Προέδρων είναι σοφή. Σήμερα ακούσαμε δήλωση του Προέδρου του Κοινοβουλίου που όπως είδα χειροκροτήθηκε από όλες τις πλευρές του σώματος. Νομίζω ότι αυτή η δήλωση είναι σημαντική και επαρκής. Τις επόμενες μέρες θα λάβουμε πολλές πληροφορίες. Θα ε, κάνουν έκτακτες συνεδριάσεις και η Επιτροπή Εξωτερικών και οι διάφορες αντιπροσωπείες. Θα δραστηριοποιηθεί και το Συμβούλιο ε, Υπουργών. Δεν θα είμαστε σε θέση να περιλάβουμε όλα αυτά τα θέματα σε ένα κείμενο το οποίο να μπορεί να τα αποκρίνεται και στην επικαιρότητα μέχρι την Πέμπτη. Δύο φορές πήγα ε, στα σύνορα της Γάζας την προηγούμενη εβδομάδα και είδα τα δεινά που ε, πάσχουν οι άνθρωποι και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Στο μέλλον δεν πρέπει να επιτραπεί πια η λαθρέα εισαγωγή όπλων στην Γάζα. Αυτό είναι σημαντικό και θα πρέπει να το λέμε. Δεν θα πρέπει οποιασδήποτε προσπάθειες γίνονται τώρα να τις ε, δυσχεράνουμε με ένα ψήφισμα το οποίο σίγουρα δεν θα μπορεί να είναι απόλυτα ισορροπημένο. Σας ευχαριστώ. Θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία με ηλεκτρονικές ε, κάρτες γιατί σίγουρα δεν θα είναι ομόφωνη. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Επαναλαμβάνω τότε. Ψηφίσατε όλοι. Αν δεν έχετε την κάρτα σας δεν μπορείτε να ψηφίσετε. Αλλά ο μόνος υπεύθυνο είστε εσείς τότε. Ψηφίσατε όλοι όσοι, έχετε τις κάρτες σας μαζί. Ρωτώ λοιπόν και πάλι. Ψήφισατε όλες και όλοι. Πέρα της ψηφοφορία. 105 υπέρ, 86 κατά. Άρα θα ψηφιστεί ψήφισμα. Κατάθεσης ε, προτάσεων ψηφισμάτων μέχρι σήμερα το βράδυ στις 8 και κοινά ψηφίσματα μέχρι Τετάρτη στις 10. Τώρα, για την Πέμπτη δεν υπάρχουν προτινόμενες αλλαγές. Ο κύριος Κον Μπέντιτ ζητεί πάλι το λόγο. Έχω μια παρατήρηση ακόμα κύριε Πρόεδρε για την συζήτηση που θα ακολουθήσει ενώ το φυσικό αέριο Ρωσία, Ουκρανία κλπ. και την σχετική... Α, ναι, είπα Σοβιετική Ένωση, συγγνώμη. <laughs> Σου ζητώ συγγνώμη αγαπητέ Βίρτς. Φρανσίς. Ε, Ζητώ συγγνώμη που αναβίωσα ένα παρελθόν, δεν το έκανα ηθελημένα. Ε, Ρωσία βεβαίως εννοούσα. Ε, διαπιστώνουμε και ελπίζουμε να συμφωνήσουν και άλλες πολιτικές ομάδες ώστε στην συζήτηση αυτή να τεθεί και το θέμα της Σλοβακίας η οποία Σλοβακία παρανόμως θέτει σε λειτουργία και πάλι πυρηνικό εργοστάσιο. Ε, ε, εσύ Φέρμπερ δεν χρειάζεται να μιλάς. Είσαι ήδη υποψήφιος στην πατρίδα σου. Αυτό ήταν όλο. Πρόεδρος, πρόεδρος. Τώρα παρακαλώ οι κύριοι Κονμπέντιτ και Φέρμπερ να πάψουν τον διάλογο. Στην συζήτηση αυτή μπορεί να συζητηθεί βεβαίως οτιδήποτε έχει σχέση με το θέμα. Έχω τώρα και μια δήλωση του κυρίου Δημητρακοπούλου. Στο πολύ κύριε Πρόεδρε. Επειδή το θέμα της σλοβακίας και της βουλγαρίας είναι σοβαρό θέλω και εγώ να σας παρακαλέσω να διαβιβάσετε στην ευρωπαϊκή επιτροπή που έτσι κι αλλιώς είναι και ο θεματοφύλακας των συνθήκων και της συνθήκης ένταξης να μας ενημερώσει για το τι ακριβώς συνέβη και γιατί πήρανε αυτή την απόφαση οι δύο αυτές χώρες. Ευχαριστώ. Είμαι βέβαιο ότι το σημείωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να το λάβει υπόψη της και μπορούμε να θεωρήσουμε λοιπόν ότι εγκρίνεται η ημερησία διάταξη. Θα έλθουμε τώρα στις ε, λήψεις λόγου για ένα λεπτό. Ο κύριος Παπαστάμκος. Επιτρέψτε μου να ενημερώσω το Σώμα για την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας κατά της Ελλάδος οι συνεχείς παραβάσεις και παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου οι χαμηλές υπερπτήσεις μαχητικών αεροπλάνων πάνω από